sind die Preisträger στα θεωρία μας, στα θεωρία τιμής συμπαρίστανται επισκέπτες σήμερα στις 17 και 30 στην αίθουσα Γεχούντι Μενουήν θα διεξαχθεί τελετή για την βράβευση των προσώπων αυτών που όπως είπα έχουν βραβευθεί με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτου. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η μερίσια διάταξη το σχέδιο των εργασιών που έχει εγκριθεί στις 11 Φεβρουαρίου από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου και το οποίο σχέδιο έχει διανεμηθεί. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ζητεί δήλωση από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη εκπρόσωπο για τα εξωτερικά ως πρώτο τελευταίο θέμα δήλωση για την κατάσταση στην Βενεζουέλα. και με ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί τον Μάρτιο στο Στρασβούργο. Επίσης το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητεί παράτηταση της σημερινής συνεδρίας μέχρι τις 10 το βράδυ. Τον λόγο λαμβάνει ο κύριος Τεγκράντης Πασκουάλ. Κύριε συνάδελφο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το αίτημα εκφράζεται σαφέστατα. Θέλουμε να τροποποιηθεί η μερίσια διάταξη και να προσθεθεί συζήτηση για τη Βενεζουέλα. Θέλουμε να υπάρξει και πρόταση ψηφίσματος η οποία να ψηφιστεί στην επόμενη ολομέλειά μας στο Στρασβούργο. Ποιοι είναι οι λόγοι. Το Δεκέμβριο το σώμα αυτό ανέκρινε ψήφισμα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία μάλιστα όσον αφορά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Έχουν περάσει τρει μήνε και η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Αντίθετα, σύμφωνα με όλα τα μέσα ενημέρωση του κόσμου, φαίνεται ότι η κατάσταση είναι έκτακτη εκεί. Διότι υπάρχουν ε, πολιτικές διώξει κατά τη αντιπολίτευση και μεγάλος ε, κίνδυνος ε, ταραχών. Νομίζω λοιπόν ότι δικαιολογείται απόλυτα το ψήφισμά μας. Ένα παιδί 12 χρονών πέθανε στα πλαίσια μια αντιπαράθεση πριν από λίγες μέρες. Γι' αυτό λοιπόν, Πρόεδρε, και ζητάμε να γίνει συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος Σούλτς. Ποιος επιθυμεί να αγορεύσει υπέρ της αιτήσεως του κ. Τέγκραντς Πασχάλου. Κανείς. Ε, ποιος επιθυμεί να αγορεύσει κατά. Κύριε Αλμπιόλ. Συγγνώμη, κύριε Αλμπιόλ. Ευχαριστώ. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά είμαστε κατά του να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Γιατί εμεί πιστεύουμε ότι ο μόνο λόγο για να συζητηθεί σήμερα στην Ολομέλεια αυτό, ο μόνο λόγο που υποβάλλεται το αίτημα αυτό να συζητηθούν όσα έγιναν ε, στο Καράκα ε, για κάποιον ο οποίο ε, εμπλέκεται σε μία υπόθεση για πραξικόπημα, πιστεύω ότι πρόκειται εδώ πέρα για πράγματα που έχουν να κάνουν με τι τροποποίησει στη Λατινική Αμερική διότι θέλετε να στηρίξετε τα σχέδια της δεξιάς κυβέρνησης και όχι όπως έγινε το 2012 με το πραξικόπημα του Τσάβες. Πρόκειται για μια κυβέρνηση που το μόνο που θέλει να κάνει τώρα είναι να βγάλει από τη φτώχεια και την πείνα εκατομμύρια ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Ο κύριος διακόπτει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος Σούλτς, περιμένετε μια στιγμή κυρία Αλβιώνα. Α, τελειώσατε, καλά. Ε, θα σας δώσω και λίγο περισσότερο χρόνο να χωρέψω, αλλά τελειώσατε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε τέτοια διαδικαστικά παρακαλείστε να ακούτε προσεκτικά μέχρι τέλους. Δεν πρόκειται να καταχραστεί κανείς της εμπιστοσύνης, της ε, υπομονής σας, συγγνώμη. Αλλά τώρα πάντως ολοκλήρωσε η κυρία Αλμπιόλ. Κυρία Αλμπιόλ, ήθελα να σας προσφέρω λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά ήσασταν ταχύτεροι. Ψηφίζεται τώρα η πρόταση του κυρίου Δεγκράντης Πασκουάλ. Παρακαλώ με έγερση του χεριού. Κατά. Αποχές. με μικρή μόλις πλειοψηφία, λέει ο Πρόεδρος, νομίζουμε χαριτολογώντας, έγινε δεκτή. Αυτό σημαίνει ότι η συνεδρίαση θα παραταθεί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ απόψε. Το πρώτο θέμα τώρα της ημερησίας διατάξεως. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα στρατηγικό σχέδιο για την Ενεργειακή Ένωση. Και δίνω το λόγο στον κύριο Μάρο Σεύκοβιτς που είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Honorable Mr. President, members. Αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, η απόφαση που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγε ώρε